αν κάποιος θέλει να τους υψώσει μπλε κάρτα να έχει έστω αυτή την ευκαιρία. Yes, yes, Mrs. Regner, you are very right. Έχετε απόλυτο δίκιο κυρία Ρέγνερ. Θα πρέπει τα μέλη να περιμένουν κάθε φορά μήπως τεθούν ερωτήσεις από τους συναδέλφους τους. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ιδίω οι άντρες, τις κυρίες. Έχετε απόλυτο δίκιο λοιπόν. Θα πρέπει τα μέλη να περιμένουν εφόσον υπάρξει ερώτηση με τη γαλάζια κάρτα. Λοιπόν, σημειώνουμε την ε, σύστασή σας και θα φροντίσουμε να συμμορφωθούμε. Συνάδελφοι, επειδή αυτή τη στιγμή επισκευάζεται το σύστημα, θα περιμένουμε λίγα δευτερόλεπτα για να αρχίσουμε τις ψηφοφορίες. Υπάρχει ένα νέο μέλος ανάμεσά μας, οπότε πρέπει να προσαρμοστεί το σύστημα και στις δικές του τις ανάγκες για να λειτουργήσει. Μόλις είναι έτοιμο, ξεκινούμε. Και τώρα θα ψηφίσουμε την έκθεση Kirkhope. Ισλανδία, Λιγνεστάιν, Ορβηγία και Ελβετία σε σχέση με το κεκτημένο Σέγγεν. Ενιαία ψηφοφορία. Μία και μόνη υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Έκθεση Μπερές. Προσανατολισμοί πολιτικών απασχόλησης. Ονομαστική ψηφοφορία ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Aprobado. Εγκρίνεται. 591 ψήφισαν υπέρ. Και πάμε τώρα. Έκθεση Αλεξάνδρ, πρώτη ανάγνωση σε σχέση με την θέση του Συμβουλίου. Ναι, κύριε Μπερές, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, θα ψηφίσουμε την έκθεση του κυρίου Σέρκας ο οποίο εξ ονόματο όλων των συναδέλφων, ιδίω της Επιτροπή Απασχόληση και Γεωργία ζητά την παράταση βάσει συμφωνία που έγινε στο Συμβούλιο του προγράμματο για την βοήθεια των μειονεκτούντων επί δύο χρόνια. Δεδομένων των πολιτικών συνθεκών εντό των οποίων συνήθει η συμφωνία αυτή στο Συμβούλιο, καταφέραμε να αποσπάσουμε δήλωση από την Επιτροπή για την δική τη. θα θέλαμε μάλλον να αποσπάσουμε μια, πρόταση, μια δήλωση από την Κομισιόν, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την δική τη θεώρηση για το μέλλον του προγράμματο αυτού. Κύριε Επίτροπε, έχετε τον λόγο. Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, κυρία Μπερές. Είμαι βέβαιος, θα γνωρίζετε, ότι το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο εγκρίθηκε στις 29 Ιουνίου 2011 και προβλέπει η μελλοντική επιστημιστική βοήθεια για τους πλέον μειονεκτούντες να χρηματοδοτείται από το κεφάλαιο 1. Εκεί συνάδει καλύτερα και με του στόχου καταπολέμηση τη φτώχεια ε, στα πλαίσια τη στρατηγική του 2020 για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν έσχισε το δικαίωμα πρωτοβουλία που έχει προκειμένου να σκεφτεί ποτέ θα υποβάλει την ανάλογη πρόταση. Το δικαίωμα πρωτοβουλία, όπω γνωρίζετε, ανήκει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πασάμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα προχωρούμε στην εξέταση τη Δευτέρα Αναγνώσεως τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά την διανομή των ε, ε τροφίμων ή σε αυτού που έχουν ε, ανάγκη. Κυρία Σικέρσκη, ε, είστε ο εισηγητή, δεν έχουμε κάποιο θέμα και επομένω εγκρίνεται η στου αυτου που εχουν αναγκη και κύριοι, ειστε ο εισηγητη Συμβουλίου. Και τώρα. Εξέταση. Δεύτερη ανάγνωση τη θέση του Συμβουλίου σε σχέση με την πολιτική του ραδιοελεκτρικού φάσματος. Έκθεση Χόκμαρκ. Τροπολόγια υπερθμών 1 με νομιστική ψηφορία ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Επομένως, εγκρίνεται η θέση του Συμβουλίου. Και τώρα, έκθεση Νίκολσον. Όσον αφορά τις συμβατικές σχέσεις εις τον γαλακτοκομικό τομέα. Πρώτα-πρώτα θα ψηφίσουμε μια, την συμβιβαστική υπαριθμόν 1. Συμβιβαστική υπαριθμόν 1. Οι δέσμοι των συμβαστικών ψηφίζεται, εγκρίνεται. Τώρα, την πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το σύνολό τη, υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε το σχέδιο του νομοθετικού ψηφίσματος με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Πέρα. Γίνεται με ευρία πλειοψηφία. Και τώρα ψηφίζουμε την έκθεση Ιλτσεφ που αφορά την τροποποίηση του άρθρου 48 του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αφορά τις εκθέσεις ιδίες πρωτοβουλίας. Απαιτείται ειδική πλειοψηφία. Τροπολογία υπαριθμών 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία παριθμών 6. Ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Πέρας. Και εγκρίνεται με την ειδική πλειοψηφία. Και τώρα. ψηφίζουμε το σχέδιο απόφασης χωρίς τροπολογίες. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έκθεση Οικονομικής Επιτροπής όσον αφορά τα ομόλογα σταθερότητος. Το πολύ υπαριθμόν ένα Υπέρ. υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται και τώρα θα ψηφίσουμε την ε, παραγραφό 4 εις δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές να εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά ε, επαλήθευση για το δεύτερο τμήμα ηλεκτρονική ψηφίζουμε Πέρας. Απερίφθη το δεύτερο τμήμα. Τώρα ψηφίζουμε. Τροπολογία παρελθόν 2. Υπέρ. Απορρίπτεται. Υπαλήθευση. Τροπολογία παρελθόν 2. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Ε, παράγραφος 9, εις δύο τμήματα. Για το πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Και το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Είναι επαλήθευση για το δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Όντως απορρίπτεται. Και τώρα. Τροπολογία υπαριθμών 3. Υπέρ. Κατά. Τροπολογία. Όχι, όχι, όχι. Διορθώνει ο πρόεδρος. Μιλούμε για τώρα για την παράγραφο 11 ε, εδάφιο 7. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλετε έλεγχο. Επαλήθευση βεβαίως. Για την ε, παραγραφό αυτήν και το εδάφιο υπερθυμών 7. 11, 7. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Ναι, εγκρίνεται. Και τώρα. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Γνωστή ψηφοφορία τώρα για την 12η παράγραφο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. το σχέδιο ψηφίσματος με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρινέται με ευρία πλειοψηφία. Έκθεση Κορνέλησεν την ε, απασχόληση και θέματα κοινωνικής πολιτικής σε σχέση με την ετησία έκθεση για την ανάπτυξη ε, ε, το 2012. Ψηφίζουμε την παραγράφο 6 εις 2 θέματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παραγραφός 7, εις τρία τμήματα θα ψηφίσουμε. Το πρώτο, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Ονομαστική ψηφοφορία. Για το δεύτερο τμήμα, ονομαστική. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα με ευρία πλειοψηφία. Τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 18. Με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται το 18. 19. Εις τρία τμήματα. Το πρώτο. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. Το τρίτο, με ονομαστική. Πέρας. Εγκρίνεται το τρίτο τμήμα. 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Σαν Ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Πέρας. Και τώρα ψηφίζουμε το σύνολο του ψηφίσματος. Υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Έκθεση. Γκοζές. Συμβολή στην ετήσια έκθεση για την ανάπτυξη του 2012 και ψηφίζουμε την τροπολή 2 υπέρ κατά απορρίπτεται. Τροπολογία υπαριθμών 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία υπαριθμών 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία υπαριθμών 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το συνοτού ψηφίσματος τώρα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πολύ καλό. Για τώρα αρχίζουμε τις επεξηγήσεις, δηλώσεις ψήφου.